Ας μην μείνουμε λοιπόν πίσω και από αυτή την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα εξαρθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ριβελίνη, περιοχή της Συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για τη Μεσόγειο. Το λόγο έχει Καταρχάς για τέσσερα λεπτά ο εισηγητής μας ο κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρούσα πρόταση κανονισμού θέλει να κάνει κάποιες συστάσεις, να εφαρμόσει από την προτάση που έκανε η ΓΕΑΜ, η Γενική Επιτροπή Αλλίας για τη Μεσόγειο, για συμβάλλει στη βελτίωση της βεβαιότητας του δικαίου και μία απλούστευση γενικά του καθεστώτος. Μέχρι τώρα οι συστάσεις που υιοθέτησε η ΓΙΑΜ έγιναν αποδεκτές από την κοινοτική νομοθεσία με, ε, προσωρινά και κάθε χρόνο γίνονται κανονισμοί για τις αληθικές δυνατότητες. Το να γίνουν μόνιμες αυτές οι συστάσεις ε, απαιτούν ένα πιο σταθερό νομικό μέσο για να ενταχθούν αυτές οι συστάσεις στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει οι συστάσεις να εφαρμοστούν μέσω νομοθετικής πράξης, όπου μπορούν να προσθεθούν και μελλοντικές συστάσεις μέσω τροποποίησεων. Όσον αφορά το περιεχόμενο των συστάσεων που υθετήθηκαν από την ΓΕΑΜ εντός του κεφαλαίου 2, τεχνικά μέτρα, της προτάσεως κανονισμού, εκεί τίθενται κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά ε, την ε, ε, την αλληλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 όσον αφορά την αδειοδότηση για αλληλευτικές δραστηριότητες και την προστασία των διαφόρων φυσικών βιοτόπων τα πλοία που μπορούν να συμμετάσχουν στην αλία χρειάζονται ειδική αλία, άδεια αλίας, που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα πίνακα που χορηγείται από, το κάτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κάτω μέλο. Όσον αφορά τον ληφτικό εξοπλισμό, η πρόταση του κανονισμού περιγράφει λεπτομερώς την ελάχιστη διάσταση του ματιού του δικτύου που χρησιμοποιείται στη Μεσόγειο, άρθρο 15, και στη Μαύρη Θάλασσα, άρθρο 16 και απαγορεύει την χρήση των συρτών ε, που έχουν σε μεγαλύτερο από χίλια μέτρα βάθος. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε, έχουμε τα ελεκτικά μέτρα. Εδώ προβλέπεται ότι κάθε κάτος μέλος διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πληροφορικής, του μέσου πληροφορικής έναν κατάλογο επικαιροποιημένο των ε, σκαφών που ξεπερνούν τα 15 μέτρα που έχουν τη σημαία του κράτους και που είναι καταχωρημένα στη χώρα αυτή και που έχουν την άδεια να αλλιεύουν στην ε, ζώνη ΓΕΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 18. Μετά, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που αφορούν ε, το κάτω φόρτωσης. Αφορά τα σκάφη τρίτων χωρών που μπορούν να υποστούν έλεγχο και επιθεωρήσεις για τις εκφορτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21. Πέραν αυτού τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν σε σκάφος τρίτης χώρας να χρησιμοποιεί τα λιμάνια τους εάν δεν έχει σημαία συμβαλωμένου μέρους της ΓΙΑΜ. Αν το σκάφος άσκησε παράνομες δραστηριότητες αλληλευτικές που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν προστατευτεί και αν δεν έχει άδεια ισχύουσα για να αλλιεύει. Άρθρο 23. Στο τέταρτο κεφάλαιο για τη συνεργασία πληροφορίες σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, εκεί προβλέπεται συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και με το γραμματέα της ΓΙΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 24 και τη διαβίβαση εκ μέρους των κρατών μελών προς τον γραμματέα της ΓΙΑΜ ε, των διαφόρων στατιστικών στοιχείων ε, αριθμό μητρώου του σκάφους, ε, χωρητικότητα, υποδύναμη κλπ. εντός προβλεπωμένων προθεσμιών. Όσον αφορά τις διατάξεις του 5ου κεφαλαίου, τελικές διατάξεις, το άρθρο 28 και πιο συγκεκριμένα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτραπή ε, μέσω συμφωνίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τροποποιεί μέσω εκορυθισών πράξεων, διατάξεις που αφορούν διάφορα στοιχεία που δεν ουσιαστικά όσον αφορά την συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν μου δίνετε άλλα δύο λεπτά, αν, είχα, αν μπορώ να έχω άλλα δύο λεπτά, μπορώ να ολοκληρώσω. Δύο λεπτά μετά μπορώ να, δύο λεπτά μετά μπορώ να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Έχετε δύο λεπτά στο τέλο. Αν θα τα χρησιμοποιήσετε τώρα, λέει ο πρόεδρο, με τα χαρά. Αλλά δεν θα δευτερολογήσετε αντί αυτή η περίπτωση, λέει ο πρόεδρο, τον κύριο Ριβελίνη. Ναι, θέλω να τα χρησιμοποιήσω τώρα τα δύο λεπτά, λέει ο κύριο Ριβελίνη. Πέραν αυτού, παρατηρείτε ότι τα συμβαλόμενα μέρη της ΓΕΑΜ ε, έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι την προθεσμία που έχει συμφωνηθεί από την ΓΙΑΜ. Η έγκαιρη λοιπόν εφαρμογή απαιτείται ούτω ώστε αυτά τα μέτρα να έχουν διεθνή χρειά και να εφαρμόζονται άμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε επίπεδο κοινοτικό και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. Όμως η διαδικασία της συναποφάσεως λόγω της μακράς διαρκείας αυτής, σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη φαίνεται ε, να είναι υπερβολική όσον αφορά τα δικαιωμένα θέματα, όσον αφορά την αποδοχή των των διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο 28, που πιστεύω ότι δεν αφορούν σημαντικά θέματα και πριν αθετηθούν στην ετήσια σύνοδο της ΓΙΑΜ, ε, ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη-μέλη και σε ομάδα εργασίας και στο Συμβούλιο και ε, στην ίδια τη Σύνοδο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται μπορεί να θεωρηθεί μια παραβίαση των διεθνών της υποχρεώσεων. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα πλαίσια της ΓΙΑΜ και άλλων διεθνών οργανισμών διαχειρίσεως της αλίας. Αυτό δεν είναι κάτι που εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα θα, χρειάζ, θα δίνει και άλλα στοιχεία σε εκείνους που είναι αντίον της Ενώσεως που μπορεί να ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση χρονοτριβή επί ασημάτων θεμάτων, δηλαδή επικεντρώνεται επί των πιο ουσιαστικών. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι σημαντικοί μηχανισμοί διαφύλαξη έχουν συμπεριληφθεί στο σύστημα των κατεξοδότηση πράξεων. Δηλαδή, η δυνατότητα προβολή αντιρρήσεων από του δύο νομοθετικέ αρχέ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των κατεξοδότηση πράξεων. Δυνατότητα να ανακληθεί επίση αυτή η εκχώρηση, αν υπάρχει ικανοποίηση για τον τρόπο με τον χρησιμοποιούνται αυτέ οι εξουσίε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι το άρθρο 28 που, αφ... μισό λεπτό, μισό λεπτό, που αφορά τι κατεξοδότητε συμπράξει, αποτελεί καλό συμβιβασμό που θα πρέπει όμω να επασυζητηθεί σε δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο, τόσο ώστε να εξευρεθεί μια οριστική συμφωνία. Αυτή η λογική ευθυγραμμίζεται με την έκθεση του κ. Μπάντε Μπρούν όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 998 που αφορά τους όρους αστυνόμευσης υγείας που, και τη διάθεση των ζώων για μη εμπορικό σκοπό. Τελειώνεται, λέει ο πρόεδρο, η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκαθιδρεί ένα πρόγραμμα τεκμηρίωση ε, τη ε, αλληλεία του ερυθρού τόνου. Θα πρέπει να μου κάνετε ένα εικόνισμα στο γραφείο σας κύριε Ριβελίνη, μπορώ να σας το βάλω και με αυτόγραφο, να έχετε φωτογραφία μου. Εν είδη για αυτά που συνέβησαν σήμερα. εγώ πάντως εικόνισμα δεν θα, δεν θα βάλω δικό σας κύριε Πρόεδρε, οπότε θα είμαι σύντομη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα όλα ευχαριστήσω τον κύριο Ριβελίνη για τη δουλειά του επί της εκθέσεως και είμαι πολύ ικανοποιημένη ε, που διαπιστώνω την στήριξη της Επιτροπής Αλληλείας ε, και του Κοινοβουλίου ε, επί της ουσίας της σημαντικής αυτής πρότασης. Εύκολα μπορώ να συμφωνήσω με την παρουσίαση του κυρίου Ριβελίνη και συμφωνώ πως η εφαρμογή των διαφόρων μέτρων που υιοθέτησε η ΓΙΑΜ είναι κλειδί στην ε, βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών πορών της Μεσογείου. Πρέπει να το κάνουμε γιατί η Μεσόγειος το χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την βιοπικιλότητα της Μεσογείου και να διασφαλίσουμε το ότι η Μεσόγειος δεν θα γίνει νεκρά θάλασσα να αναφερθώ σε ένα θεσμικό ζήτημα που ανέφερε και ο κύριος Ριβελίνη. Όπως ξέρετε, οι συστάσεις της ΓΙΑΜ γίνονται δεσμευτικές επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα στα κράτη-μέλη από τη μέρα που ορίζεται από την ΓΙΑΜ. Οπότε η έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για έτσι ώστε τα διεθνή αυτά μέτρα να έχουν άμεση ισχύ επιφυσικών ή νομικών προσώπων και να υπάρχει νομική ασφάλεια. Οπότε, αγαπητοί βουλευτές, πρέπει να αποφύγουμε το, η εφαρμογή των μέτρων της ΓΙΑΜ να γίνει ε, μια συσύφια υπόθεση. Ήδη τώρα η μεταφορά τέτοιων μέτρων που υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια ο ΓΕΑΜ εκρεμεί λόγω μη υιοθέτηση του κανονισμού. Αλλά σύντομα ο ΓΕΑΜ θα υιοθετήσει πιθανότατα νέες τροποποιήσεις που απαιτούν αποτελεσματική ε, μεταφορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Οπότε κάνουμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Γι' αυτό θεωρώ πως η Επιτροπή θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες εξουσιοδότηση για να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο όλες οι μελλοντικέ τροποποιήσεις. Γιατί ενισχώ πως εάν δεν γίνει αυτό θα έχουμε υψηλούς κινδύνους μη έγκαιρης μεταφοράς αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Δεν είναι αυτός ένας τρόπος ε, να αποφύγουμε την αρποδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά χρειάζεται έγκαιρη μεταφορά στο δίκαιο και φοβάμαι πως μέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα γίνει κάτι τέτοιο δυνατόν. Γι' αυτό λυπούμε για το ότι δεν συμφωνούν τα θεσμικά όργανα και θα ήθελα να τονίσω πως οι καθυστερήσεις αυτές θα καθυστερήσουν την δυνατότητα της Ένωσης να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, θα υποβαθμίσουν την ε, αξιοπιστία μας ε, στους διεθνείς οργανισμούς αλληλείας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θεωρώ πως θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την υιοθέτηση αυτού του οργανισμού γρήγορα και άρα καλωσορίζω την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω πως περαιτέρω παρόμοια βήματα θα μας επιτρέψουν να ξεμπλοκάρουμε τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση της πρότασης ταυτόχρονα. Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς στο, εθνικό, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέτρων από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης αλίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητούμε καλύτερες λύσεις και σας ζητώ να συνταχθείτε μαζί μας. Οπότε πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ριβελίνη για την έκθεση και την Επιτροπή της Αλληλείας για τις προσπάθειές της. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you, Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος ε, Κάρτεκ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω καταρχάς ότι Είμαστε εδώ στο Στρασβούργο. Είμαστε ωραία εδώ στο Στρασβούργο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ριβελίνη ε, για την εκθεσή του και για τη συνεργασία του ε, από το 2009 και με μια περίοδο που είχαμε κάποια αναστολή κάποιων πράξεων ε, με τη συνδίκη της Αβώνας κτλ. Τώρα στην έκθεση αυτή μεταφέρονται κάποιες διατάξεις που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση σύσταση η οποία έχει ε, υιοθετηθεί από τη ΓΙΑΜ ουσιαστικά επιβάλλει κάποιες ε, περιορισμούς σε ό,τι αφορά τα μάτια των δικτυών, σε ό,τι αφορά τα ενδιατήματα και είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει κάποιες αληφτικές ζώνες ε, στη Μεσόγειο. Το κείμενο περιγράφει λοιπόν το κατώτατο, τις κατώτατες της διατάξης των ματιών και στην Μαύρη Θάλασσα και στην Μεσόγειο και επίσης απαγορεύει τη χρήση σειρώμενης δράγας και τράτας σε βάθος ανώτερο των χιλιών μέτρων, κάτι που θέλω να το επικροτήσω. Θα πρέπει λοιπόν είτε να έχουμε 40 εκατοστά ε, μάλλον 40 mm στο ανώτερο μέρος του σάκου στο δείχνει με τετράγωνα μάτια ή να έχουμε ρομβοειδή μάτια 50 ε, mm. Ε, με επιστοποιημένη επιλεκτικότητα αναλόγως του μεγέθους, ισοδύναμη μεγαλύτερη των δικτυών με τα τετράγωνα μάτια. Θα πρέπει επίσης να Είμαστε πολύ ξεκάθαροι και στην ε, θέση την οποία θα υιοθετήσουμε και θα τα πω και στην κυρία Επίτοπο. Θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 να έχει υποβληθεί έκθεση για την ε, υλοποίηση μεταφορά στο Εθνικό ε, Δίκτυο και θα πρέπει να, δίκαιο και θα πρέπει να υπάρξουν ίσως και κάποιες προσαρμογές. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του κειμένου. Ευχαριστώ. Thank you very much Mr. Arsenis. Ευχαριστώ κύριο για δύο λεπτά. Πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι η μεσόγειος αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι του πλανήτη μας μόλις το 1% περίπου της θαλάσσιας περιοχής όμως είναι πάρα πολύ πλούσια έχει το 8 με 9% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 50% των αλλιευτικών σκαφών της Ευρώπης βρίσκονται στη Μεσόγειο 60% ε, της εργασίας, της απασχόλησης στην αλληλεία λαμβάνει χώρα στη Μεσόγειο αλλά δυστυχώς το 54% των ε, αλλιευμάτων υπεραλλιεύεται. 32 με 36% των αλλιευμάτων βρίσκονται εκτός βιολογικών ορίων. Τι φταίει, προφανώς η αποτυχία της έως σήμερα κοινή αλλιευτικής πολιτικής, η μη εφαρμογή πολλές φορές των κοινών μας αποφάσεων, αλλά κυρίως και αποφάσεις που λαμβάνουμε χωρίς να σεβόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα, αποφάσεις που λαμβάνουμε κινούμενοι από κακώς νοούμενα εθνικά συμφέροντα. Το 2006 η Επιτροπή προσπάθησε να διορθώσει τα προβλήματα της Μεσογείου. Είχαμε την, ε, το κανονισμό της, ε, για την αλληλεία στη Μεσόγειο, όμως τα προβλήματα δεν σταματάνε μόνο στο τι κάνουμε εμείς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεία στη Μεσόγειο και το μέλλον των αλληλευμάτων εξαρτάται από το τι κάνουμε όλες οι μεσογειακές χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι σε αυτό το κοινό μας πλούτο. Και αν δεν δράσουμε από κοινού, ο κοινό μας πλούτος αυτός κινδυνεύει άμεσα προχωρήσαμε στην ε, πρώτη ανάγνωση ε, της έκθεσης αυτής. Με λύπη το Συμβούλιο το οποίο απουσιάζει και σήμερα από αυτή την αίθουσα ε, είχε μια ακατανόητη αιμονή στα θέματα της πρόθεσης των μέτρων εφαρμογής, των Implemented measures. Το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβει ότι η συνθήκη Λισαβόνας πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να δεχθεί το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει στις αποφάσεις αυτές και να δεχτεί τα μέτρα κατευσιοδότηση, τα delegated acts. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα έχει Ευχαριστώ. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες εφαρμογής της κοινή εθνικής πολιτικής έδωσαν ότι θα πρέπει να θεσπιστεί δεν εφαρμόζουν σωστά μέτρα στη διαχείριση της αλίας στην Ευρώπη. Έχουμε πόλεμο Ατλαντικού κατά Μεσογείου. Οπότε έχουμε ένα ε, κακή διαχείριση σε status quo. Δεν εφαρμόζονται τα μέτρα και υπάρχει υπεραλίευση στη Μεσόγειο. Μόνο οι αλληλείς και οι κυβερνήσεις, αν γίνουν υπόλογοι της Μεσογείου και εργαστούν με τις χώρες του Ατλαντικού και εφαρμόζουν κοινέ διαδικασίες και μέτρα, μόνο τότε μπορούμε να φύγουμε από το παρελθόν, να ξεφύγουμε ούτε τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου και τα λιεύματα, ούτε οι αλληλείς μπορούν να αποδεχτούν νέα αποτυχία της κινησερευτικής πολιτικής αυτή τη φορά όσον αφορά τη Μεσόγειο. Η αλληλεία στη Μεσόγειο πρέπει να καλύπτεται σωστά, να καλύπτονται όλες οι πτυχές της από τη νέα αλληλευτική πολιτική, να καλύπτεται η Μεσόγειος. Δηλαδή τα μέτρα διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζονται Χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αλληλευτική προσπάθεια και τη διαχείριση αυτής στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες προδιαγραφές όπως τα μέτρα που εφαρμόζονται και την αλληλεία στη Μεσόγειο. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ Ατλαντικού και Μεσογείου. Ευχαριστώ. κύριος Φόξ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, την κυρία Δαμανάκη για την πρότασή της για να σταματήσει η αποκρουστική αυτή πρακτική της απόρριψης. Όταν μειώνονται τα αποθέματα και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αφάνε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι κρίμα να πιάνουμε μια χαραψάρια, τα σκοτώνουμε και να τα ξαναπατάμε στη θάλασσα για να ταΐζουμε τους γκλάρους. Ελπίζω λοιπόν να εφαρμοστεί άμεσα η νομοθεσία για να σταματήσει αυτή η επέσχυντη πρακτική των συντομότερων δυνατών πέραν από την πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν καλωσορίζω και τις στάσεις του ΓΕΑΜ. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τις προτάσεις όσον αφορά τον ελευτικό εξοπλισμό και του ελάχιστου μεγέθους ματιού για την ε, Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγεια και την απαγόρευση ε, των ε, παρασυρωμένων δικτυών κάτω από το όριο των χιλίων μέτρων. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Δαμανάκη προσωπικά για την κατάργηση των απορρίψεων. Ευχαριστώ κύριε Βαλένζα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να τονίσουμε πως η Μεσόγειος είναι η μόνη θάλασσα στον κόσμο που περικλείεται από τρεις υπήρους με πολλούς πολιτισμούς και πολλές τρίτες χώρες επίσης. Οπότε το, τα βασικά ζητήματα όσον αφορά την ε, θαλάσσια οικονομία της Ένωσης είναι η ρύθμιση της αλληλείας αλλά οπωσδήποτε και η ανάπτυξη ε, μέσων εποπτείας ε, των λευτικών σκαφών που δρούν εκεί πέρα. Οι αλληλοί στη Μεσόγειο βεβαίω απολαμβάνουν τον πλούτο των ειδών εκεί πέρα. Οπότε για να υπάρχει δίκαιη εκμετάλλευση της θάλασσα αυτής χρειαζόμαστε μέτρα όπως αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ριβελίνη για την ικανότατη αυτή έκθεση η οποία ορίζει τρόπους διαχείρισης των πόρων ε, της Μεσογείου που είναι πολύ πολύτιμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριος Μιλάνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ε. Θεωρώ ότι τα θέματα που σχετίζονται με τη Μεσόγειο, με την διάταξη αυτή, ξεκινούν μια φάση πολύ πιο σημαντική από τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τούδε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντική η πράξη που συζητάμε σήμερα με, από τις επιπτώσεις του κανονισμού του 2006 θεωρώ ότι αυτό απαντά και στους περιορισμούς που είχε ο συγκεκριμένος κανονισμός, διότι είχε αφήσει πολλές φορές ε, τομείς αλληλείας ε, οι οποίοι πίστευαν ότι η Ευρώπη κάνει όσα πρέπει να κάνει αλλά τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου δεν το κάνουν. Είναι, πολύ είναι στρατηγική σημασία για μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα λοιπόν σε αυτές τις διαστάσεις και με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα όσα έκανε ο κύριος Ριβελίνη είναι ε, στοιχεία με τα οποία συμφωνώ και εγώ και νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε επισήμω εδώ. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι εμείς δεν καταφέρνουμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση και θα καταλήξουμε τελικώς σε δεύτερη ανάγνωση, κυρίως για την ερμηνεία του άρθρου 28 του συγκεκριμένου κανονισμού, θέτει ένα ερωτηματικό. Το Κοινοβούλιο ε, σε αυτή την περίπτωση τάσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο λέει ουσιαστικά ότι είναι καλό αυτές οι πράξεις εξουσιοδότηση να υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αντιτίθεται και μάλιστα η σημερινή του απουσία είναι προφανής για το θέμα αυτό. Στο Κοινοβούλιο έχει οριμάσει η άποψη ότι το να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα, το να διατηρήσουμε τη δυνατότητα αλίευσης αυτής της τόσο σημαντικής θάλασσας είναι το μέλλον των αλλιέων. Πέραν αυτού όμως, εγώ θεωρώ ότι η φάση που έχουμε ενώπιόν μας θα πρέπει να διατηρήσει στο επίκεντρο την ιδέα της συναπόφασης. Αυτές οι πράξεις κατεξουσιοδότησης έχουν λόγο για τον οποίο εξουσιοδοτούνται και θέλουμε να τα εξουσιοδοτήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι συμφωνίες όταν θα γίνουν θα πρέπει να διατηρήσουν σαφώς και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Χίγγινς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή Αλίας. Χαίρομαι μπορώ να υποστηρίξω αυτή την, ε, την έκθεση και οπωσδήποτε θα την υπερψηφίσω. Το 1994 όταν είχε ξεκινήσει όλη η υπόθεση επίσης ε, την υποστήριξα. Και θέλω βεβαίω να ευχαριστήσω και την κυρία Επίτροπο που απαγόρευσε τι απορρίψει πολιτικών μέτρων και σα ευχαριστούμε. Δεύτερον, για το ζήτημα τη Μεσογείου και τη ε, Μαύρη ε, Θάλασσα. Έχουμε πραγματικά έναν περιβαλλοντικό παράδεισο. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι να συγκεράσουμε όλα τα σημαντικά στοιχεία, διαχείριση, εκμετάλλευση, διαφύλαξη, εμπορία και μέτρα επιβολής, γιατί βεβαίως είναι σημαντική αυτή από την πλευρά της ιχθυοκαλλιέργειας και των προϊόντων της. Βάλαμε λοιπόν όλα αυτά τα διάφορα στοιχεία μαζί, γιατί είχαμε ξεχωριστά ψηφίσματα και κανόνες, αλλά τα φέραμε σε ένα συνολικό και λογικό πακέτο με χαρακτηριστικά πρώτα απ' όλα τη Αθήνια και δεύτερον την απλοποίηση για να καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται. Και ελπίζω αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα, υιοθετώντα αυτή την ε, έκθεση, είναι να έχουμε ένα απλοποιημένο λειτουργικό πλαίσιο για την Μεσόγειο και στο μέλλον για τη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία και στη και έχουμε τρει ομιλητέ, ξεκινώντα με την κυρία Ματέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με τον εισηγητή ω προ την ανάγκη να πλουστεύσουμε την νομοθεσία σε θέματα λία με ένα κανονισμό ο οποίο θα μπορέσει να συμπεριλάβει τι συστάσει που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αλία για τη Μεσόγειο. Συμφωνώ με τους στόχους και τις αρχές που εφαρμόζονται στην κοινή ε, αλλιευτική πολιτική, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει όλα τα παράκτια κράτη-μέλη να έχουν τη δέουσα ισορροπία μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών αξιών και διατήρηση των οικοσυστημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για την προστασία των συγκεκριμένων συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων. Ο κανονισμός αυτός επιβάλλει ελεπτομερώς ε, ε, τα εργαλεία που ε, χρησιμοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου. Να σας πω ότι ο ρόλος της διαφύριαξης των φυσικών οικοτόπων έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για κάποιες κοινότητες αλλιέων. Η Ιταλία είναι εν αναμονή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια παρέκκληση για την απαγόρευση αλληλεία δύο συγκεκριμένων ειδών που αποτελούν το βασικό προϊόν αλληλεία ε, μια συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συντονίσουμε όλους τους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θεωρεί, προσπαθήσουμε να μην είναι τόσο αυστηρά αυτά τα μέσα διότι υπάρχουν δυσκολίες επιβίωσης ε, για τις τοπικές ε, ηχθειοαλλιευτικές κοινότητες. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία τα είπατε μεν, αλλά μιλήσατε για ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα κυρία Μάτερα. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Πατράο Νέβες. Για ένα λεπτό. Um Η παρούσα πρόταση κανονισμού στόχο έχει να τροποποιήσει τις βασικές συστάσεις που έχουμε για την αλληλεία σε ένα και μόνο κανονισμό για να βελτιστοποιήσουμε τη διαχείριση και να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι συμμετέχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Οι συγκεκριμένες οικολογικές συνθήκες αυτών των ε, αποθεμάτων είναι ο βασικός ε, στόχος. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον, ε, ε, τους οικοτόπους της Μεσογείου θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση της αλίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία από τις βασικές προσκλήσεις είναι η καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Οι προτάσεις που γίνονται στο κείμενο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θετικές. Θα πρέπει ε, να γίνεται Έλεγχο όμως τη σωστή εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και όχι μόνο για το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ σκαφών ε, που πλέουν με σημαία κρατών της Μεσογείου, αλλά και ε, για σκάφη με άλλες σημαίε, με σημαίε τρίτων χωρών. Έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που αναφέρουμε για να έχουμε και ίση μεταχείριση για όλους τους στόλους που αποτελούν ε, τμήμα του αλευτικού στόλου της Μεσογείου. Ο κύριος Φερέρα για ένα λεπτό. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πτυχή αυτή τη πρόταση κανονισμού που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Δεν πρόκειται για τη συμφωνία πολυμερούς ε, συνεργασίες όσον αφορά τη διατέρηση των ε, θαλασσιών πόρων των αντίων. Η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να διευρύνει τις αρμοδιότητες κατά τέτοιο τρόπο ούτω ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ε, κρατών μέλων, παραδείγματος χάρη της Κύπρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι υπάρχουν προβλήματα με μια τρίτη χώρα που είναι υποψήφια. Κατόπιν παρεμβαίνει η πρόταση αυτή στα δικαιώματα διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων μιας χώρας. Ε, αυτό είναι όμως ένα δικαίωμα που τους δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς απαιτούμε η πρόταση που έχουμε υποβάλει να γίνει δεκτή. Δηλαδή το πεδίο εφαρμογής των πράξεων αυτών να περιοριστεί και να ψηφιστούν ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπος έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να κάνω δύο σύνομες παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με εκείνους τους βουλευτές που τόνισαν ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια καλή εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Ο κανονισμός αυτός ε, ισχύει εδώ και λίγο χρονικό ε, διάστημα. Θα πρέπει να του δώσουμε τις δυνατότητες να επιτύχει. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βελτιώσουμε ή να έχουμε περισσότερες ε, εξαιρέσεις. Υπάρχει πάρα πολύ ευελιξία θα έλεγα. Τα κρατη θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν τους κανόνες εάν θέλουν και αποκλήσεις. Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και συμφωνώ με τους βουλευτές που το ανέφεραν χρειαζόμαστε λέω στην Μεσόγειο να έχουμε μια κατάσταση παρόμοια όπως με κίνηση άλλες θάλασσες. Η Μεσόγειος χρειάζεται διακανονισμό. Είναι ανθεσφυβήτητο. Και γι' αυτό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής ελευθερικής πολιτικής θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, ούτω ώστε να έχουμε το ίδιο καθεστώς στη Μεσόδιο όπως έχουμε και σε άλλες θάλασσες της Ευρώπης. Και μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε. Η ιδέα της Κομισιόν να υπάρχουν αυτές οι ε, συμπληρωματικές πράξεις για την εφαρμογή των αποφάσεων των διεθνών σωμάτων δεν ε, ε, έχουν πει έκπτωση στην ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Τουναντίον αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει δυνατότητα διευκόλυνσης της εφαρμογής των νόμων σε ευρωπαϊκό νόμο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δαμενάκη. Κλείνει η συζήτηση. Συμφωνία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. The... Περνάμε τώρα την ερώτηση προς την Επιτροπή για την ε, Συμφωνία Ελευθερικής Συμμεταξής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της